Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι χαρά για μένα να κηρύξω την έναξη συνεδρίαση αυτή τη Επιτροπή μα, οίκων και τη Επιτροπή Προπολογισμών μαζί. Θα συνεργαστούμε σε πολύ σημαντικά θέματα. Καλή επιλογή αυτή τη διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών διότι έχουμε πολύ καλή εμπειρία συνεργασίας όσον αφορά και σε άλλες εκθέσεις ο συνδυασμός των δύο επιτροπών είναι θετικότατος. Χαρά για μένα ζω να συμπροεδρεύω μαζί σου. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 20ης Νοεμβρίου του 2017. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ε, Ευτυχώ δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Ζαν, λοιπόν, θες να αναλάβεις την Προεδρία. Χαίρομαι για μια νέα συνεργασία μεταξύ ΕΚΟΝ και Μπότζ. Έχω έξοχες αναμνήσεις από αυτές τις συνεργασίες μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο τώρα στον Επίτροπο, τον κύριο Καϊτάνεν, να μας παρουσιάσει το σχέδιο του που εμπνέεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Invest EU Program. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι πρόεδροι, συμπρόεδροι, ευχαριστώ για την πρόσκληση Μου φαίνεται σαν να συζητάμε το εύση. Βλέπω τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πρόσωπα. Αυτό είναι καλό σημάδι. Παρόλο που δεν είναι δικό μας καθήκον να επιλέγουμε συγγητές και σκιώδεις, ελπίζω όμως ότι πλανάτε γνώσεις που διευκολύνει τα πράγματα. Για το ταμείο αυτό, Invest EU Fund, τέλος 2014 ανέλαβε αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε μειωθεί κατά 15% οι επενδύσεις. Αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτική κρίση. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη ήταν συλλογική απάντηση και ανταπόκριση στην κατάσταση. Χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον εκείνων που πόλεμησαν σκληρά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στατηγικές επενδύσει. και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλου σα ε, για την καλή δουλειά που κάνατε. Παρακολουθήσατε εκ του σύνεγγυς την όλη εξέλιξή του, θα επαναλάβω τα στοιχεία. Τα στοιχεία ήδη τα γνωρίζετε. Να αναφέρω όμως κάποια υπέροχα επιτεύγματα παρόλα αυτά. Χάρη στο ΕΦΣΥ, πάνω από 640.000 μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Περίπου 15 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν ευρυζωνικό διαδίκτυο, 13.000 ΜΒ παραπάνω ε, ηλεκτρικής ενέργειας ε, παράγονται 95% από αυτό προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν από ασφαλέστερο και καλύτερο πόσιμο είδωρ χάρη στην αναβάθμιση σωλήνωση και των διαφόρων δικτύων σωλήνωση. Τα στοιχεία τι δείχνουν ότι το ΕΦΣΥ κάνει τεράστια διαφορά Σήμερα οι συνθήκες οι επενδυτικές στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί χάρη σε μεταρρυθμίσεις για την εμβάθυνση νέας αγοράς και θετικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη. Επίσης έχουν εν γέννη πιο ευνοϊκή οικονομική κατάσταση, αλλά αυτό δεν αρκεί δεν αρκεί για να αντισταθμίσει ε, έτη πολλά με πολύ χαμηλές επενδύσεις, ούτε να χρηματοδοτηθούν ανάγκες σε βασικούς τομείς όπως είναι η κυκλική οικονομία, η ψηφιοποίηση, η καινοτομία, ή κοινωνικές υποδομές και οι δεξιότητες. Δεν αρκεί να προετοιμαστούμε για τις μελλοντικές προκλήσεις. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ε, ετοιμάσει ένα εργαλείο, ε, το InvestEU Fund, που θέλει να καλύψει πολλά είδη επενδύσεων. Βασισμένοι στις ε, επιτυχίες του ΕΦΣΥ θα κινητοποιήσουμε το, με το EU Investment Fund ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις από το προπολογισμό που είναι 38 δις ευρώ για να στηρίξουμε επενδύσεις που θα εφαρμόσουμε μαζί με τους εταίρους μας και θα αυξήσουμε και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε κινδύνους. Θα πρέπει να οδηγήσει σε άλλα 650 δισεκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικέ ε, περαιτέρω επενδύσει. Το βασικό μήνυμα ποιο είναι, ότι το InvestEU ξεπερνάει το FC 3,0 για τρει λόγους. Το InvestEU είναι μεγάλη απλούστευση σε σχέση με το παρόν πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει όλη την υποστήριξη που παρέχεται μέσω 13 κεντρικά διαχειριζομένων οικονομικών μέσων και του ΕΦΣΥ σε ένα εργαλείο με πολλές πολιτικές Επίση, 13 συμβουλευτικέ υπηρεσίε θα ενταχθούν σε μία ενιαία υπηρεσία. Όλη η χρηματοδότηση και όλη η συμβουλευτική υποστήριξη εντάσσεται μέσα, από Invest, μέσα στο InvestEU, που φεύγουμε τον κατακαιρματισμό, αλληλεπικαλύψει και διευκολύνεται η ζωή για του δικαιούχου. Έτσι δε περαιτέρω θα μα επιτρέψει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα, χρησιμοποιώντα ε, λιγότερο, χαμηλότερο προπολογισμό συγκριτικά μαζεύουμε όλα τα εφιστάμενα μέσα και μπορούμε να πετύχουμε 15% περισσότερες επενδύσεις με αυτόν τον τρόπο. Το InvestEU Fund επιτρέπει επίσης πιο ομαλό συνδυασμό με τις χορηγίες και τις δωρεές. Αναμειγνύοντας δωρεές από άλλα προγράμματα όπως το Horizon Europe, το πρόγραμμα την Ενία αγορά ή το Connecting Europe Facility με υποστήριξη από το InvestEU, όλα αυτά μαζί Μέσω των κανόνων του InvestEU θα εφαρμόζονται τα προγράμματα. Δεν θα έχουμε πλέον διπλή υποβολή αναφορών, ούτε πλέον διπλέ διπλές ομάδες κανόνων. Σημαντικότατη απλούστευση. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα. Το InvestEU ε, θα καθοδηγείται προς βασικές πολιτικές. Και αυτό είναι το νέο επενδυτικό περιβάλλον. Είναι η όγκη και το μέγεθος των ποσών είναι σημαντικό, αλλά οι πολιτικές περισσότερο. Βασικός στόχος του ΕΦΣΙ είναι να κινητοποιήσει όγκο και να οδηγήσει επενδύσεις αμέσως μετά τις κρίσεις. Το InvestEU θα εδράζεται περισσότερο επί των φιλόδοξων προτεραιοτήτων των νέων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φαίνεται και στη δομή που θα έχει με την κατανομή σε τέσσερις ε, θηρίδες πολιτικής αν θέλετε. Πρώτα θέλουμε βιώσιμες υποδομές, δεύτερο θέλουμε έρευνα και καινοτομία και ψηφιοποίηση, τρίτον θέλουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καλύπτονται και τέταρτον κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Το InvestEU Fund ανοίγει και άλλες δυνατότητες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ισχυροποιήσουν επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής μέσω ε, τμήματων που αποφασίζει το κράτος μέλος. Και μπορεί να συμβάλλει το κράτος μέλος μέχρι 5% από τα ταμεία συνοχής στο InvestEU. Έτσι τα κράτη-μέλη θα ωφεληθούν από μεγαλύτερη βαθμολόγηση πιστοληψίας, οπότε θα είναι πιο ε, βιώσιμες οι επενδύσεις. Τρίτον, θέλω να πω ότι το InvestEU θα βασίζεται επί όλης της διαθέσιμης ε, τεχνογνωσίας από διάφορους εταίρους. Θα πολλαπλασιάζονται έτσι τα αποτελέσματα επιτόπου από τις επενδύσεις. Βασικός εταίρος θα παραμείνει το ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η τράπεζα θα δώσει περίπου 75% από τις εγγύησεις αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ιδιαίτεροι τομεί και γεωγραφικέ περιοχέ μπορεί να ωφεληθούν από παρεμβάσει συγκεκριμένων φορέων, όπω είναι το EPRD, το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και οι Εθνικέ Τράπεζε για Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ποια είναι η ιδέα να συνδυάσουμε την ισχύ της ομάδας ε, ε, ERB και με τη τεχνογνωσία άλλων φορέων για να κάνουμε περισσότερα, να καλύψουμε ευρύτερε περιοχέ και να καλύψουμε όμω και μικρότερα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξη. Οπότε θα έχουμε για συγκεκριμένου τομεί συγκεκριμένα χρηματοστατικά προϊόντα, για συγκεκριμένου στόχου. Λοιπόν, τώρα ποιε είναι οι τρει ομοιότητε ε, μεταξύ ΕΦΣΙ και InvestEU. Πρώτα απ' όλα βασιζόμαστε τεχνογνωσία των διαφόρων εταίρων μα ε, στον κύκλο των προγραμμάτων. Ε, θα, θα συνεργάζονται οι εταίροι και θα εφαρμόζουν και την αρχή της χρηστής διαχείρισης ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμβατότητα που υπάρχει στα, μεταξύ προγραμμάτων και πολιτικών Ευρωπαϊκό ονάσεω και ομάδα εμπειρογνωμόνων από του εφαρμοστικού εταίρου ε, ε, βαθμολογούν το πρόγραμμα και εξασφαλίζουν ότι υπάρχει ομοιόμορφη προσέγγιση. Μετά θα υπάρχει μια επιτροπή επενδυτική ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων τη αγορά που θα αποφασίζει για τη χρήση ε, των εγγυήσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Εξασφαλίζεται έτσι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα το InvestEU θα διατηρήσει βέβαια τις βελτιώσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία που εισήχθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο fc 2.1 ε, με τη δημοσίευση συστήματος βαθμονόμησης ε, και διαφόρων αποφάσεων των επενδυτικών επιτροπών. Η τρίτη ομοιότης είναι ότι υπάρχει επίσης και συμβουλευτικός φορέας και εδώ προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις. Αυτός ο κόμβος θα αντικαταστήσει 13 συμβουλευτικέ υπηρεσίε, ο κεντρικό κόμβο. Και αυτό ο κόμβο θα γίνει ένα ενίο σημείο ε, εισόδου για όλα τα αιτήματα ε, ε, ενίσχυση. Και η πύλη θα συγκεντρώνει του επενδυτέ και αυτού που εφαρμόζουν τα προγράμματα μέσω και όλοι θα εντάσσονται σε ένα κοινό τομέα δραστηριότητα. Όλοι οι φορεί που εφαρμόζουν τα προγράμματα. Συνοψίζοντα λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω τα εξή. Η πρόταση InvestEU βασίζεται στα ισχυρά σημεία του επενδυτικού σχεδίου ε, για την Ευρώπη και η συνεργασία μας μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχυροποιείται. Αλλά από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο μαθαίνουμε τα μαθήματα και έχουμε συγκεκριμένο εργαλείο που το διαθέτουμε στο οικονομικό πλαίσιο για να έχουμε επενδύσει για να πετύχουμε τι βασικέ μα προτεραιότητε. Το InvestEU θα επιφέρει απλούστευση με ένα ενιαίο εργαλείο και ενιαίο σύνολο κανόνων αντί να έχουμε πολύπλοκα διακλειδούμενα μέσα. Και είναι μια πλήρης ε, προσέγγιση που καλύπτει πολλούς με την ομάδα ε, της Ευρωπαϊκής Τάπεζας Επενδύσεων και άλλους εταίρους που μπορούν να κάνουν ε, καλύτερα τα πράγματα με μεγαλύτερη κάλυψη. Αυτά ήθελα να σας πω αγαπητά μέλη. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το InvestEU Ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία ε, και η καλή συνεργασία να συνεχιστεί όπως ήδη μέχρι τώρα κάναμε και έχουμε δείξει ότι φέρνουμε αποτελέσματα όταν το κάναμε αυτό και αποφασίσαμε από κοινό για το ΕΦΣΥ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε για αυτή την παρουσίαση. Όλο αυτό το εγχείρημα που σκοπεύει να προστεύσει τις διαδικασίες με πολλαπλασιασμό των πόρων. Εδώ έχουμε προσκαλέσει τους συνεισηγητές, πέντε λεπτά για τον καθένα και κύριε Αντιπρόεδρε, μετά τις παρεμβάσεις τους θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε. Μετά θα δώσουμε το λόγο στους και όντες εισηγητές, δύο λεπτά στον καθένα. Και για να γίνει πιο ζωντανός ο διάλογός μας θα απαντάτε σε κάθε ερώτηση κύριε Επίτροπε. Ο λόγος στον κύριο Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για αυτήν την κοινή συνετρίαση. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά μαζί και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για την προσελευσή του. Ελπίζω όλη αυτή δουλειά που έχει προηγηθεί να γίνει επιτυχημένη ιστορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες και να στηρίξει την οικονομία. Δεν άκουσα τον όρο προσθετικότητα. Στο ΕΦΣΙ πρώτη έκδοση και δεύτερη έκδοση μόνο αυτό ακούγαμε. Σορευτικότητα, προσθετικότητα. Εάν το κριτήριο αυτό θα ε, συνεχίσει να υπάρχει όχι, δεν το ξέρουμε. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε σχέση με την ανάγκη τη της... της προσθετικότητας. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι προσφέρουμε βεβαιότητα και δυνατότητα να είναι τα πράγματα προβλέψιμα. Πώς θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υπάρχει αυθαιρεσία ή τέτοια διακριτική ευχαίρεια που να καταλήγει να γίνεται αυθαιρεσία. Και να μην παίρνουμε χρήματα και πόρους από ένα χρηματοδοτικό μέσο για να τα πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή ευελιξία να υπάρχει, αλλά να υπάρχει και δυνατότητα προβλεψιμότητας. Επίσης, Ε, επίσης για την ε, εδαφική συνοχή το ταμείο αυτό δεν είναι ταμείο συνοχής αλλά δεν θέλουμε να αντίκειται και στις προσπάθειες της συνοχής και εδώ με ενδιαφέρει και η γεωγραφική κατανομή και θεματική κατανομή πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει τον στόχο να υπάρχει αυτή η γεωγραφική κατανομή μια τέτοια κατανομή που να είναι και ε, σωστά εξισορροπημένη. Βεβαίως υπάρχουν εδώ ε, αντίρροπες δυνάμεις, ε, δυνάμεις αποκέντρωσης. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε και ελπίζω να ενισχυθεί και αυτό το hub το συμβουλευτικό, αυτό το κέντρο το συμβουλευτικό για να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Κάτι ακόμα είναι οι εγγυήσει και οι χρηματοοικονομικές τράπεζες ανάπτυξης των κρατών μελών ποιο μέρος θα πηγαίνει στην ΕΤΕ ως προς την εγγύηση και ποια θα πηγαίνει στις επενδυτικές τράπεζες των κρατών μελών ή τέλος πάντων στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ανάπτυξης των κρατών μελών. Ε, και μία ακόμη ερώτηση. Πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ άλλα ε, ε, έχουν αδύναμα τέτοια ιδρύματα. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι θα ληφθεί αυτό υπόψη. Στο ΕΦΣΙ 2 τα ε, όμορα κράτη μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση. Αυτός ο όρος διατηρείται. Πώς μπορούμε να καταρτήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα που το InvestEU να μπορεί να συνδεθεί και με παρόμοια ταμεία ή καταπιστεύματα όπως αυτό της Αφρικής ε, ή αυτό της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ή το Ευρωκοινοβούλιο είχε δίκιο όταν έλεγε ότι 40% για το Ταμείο των Αγγίσεων ήταν ε, αρκετό. Ήταν αρκετό για να συγκροτηθεί ταμείο, να συσταθεί. Ε, κάτι ακόμη που βλέπω είναι ότι είναι 13,7 και όχι 15 ο συντελεστής πολλαπλασιασμού. Ποια ε, η σχέση λοιπόν με τα διευθυντικά ταμεία, πώς θα υπάρξει αλληλεπίδραση. Εγώ θεωρώ θετικό το γεγονός να υπάρχει δυνατότητα το InvestEU να χρησιμοποιείται ανά κράτο μέλο, ώστε το 7% των ε, εθνικών χαρτοφυλακίων να πηγαίνουν και να κινητοποιούν επενδύσεις. Είναι ένας ε, τρόπο να μπορούμε να παρακάμψουμε το πρόβλημα του να μην υπάρχει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που να είναι αρκετά ε, σταθερό, ε, αρκετά ισχυρό. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν σωστά αυτή η μετάβαση, το 7% βεβαίως, είναι κάτι που προβλέπεται σε θελοντική βάση. Αλλά γιατί 7 και όχι 6 ή κάτι άλλο. Αυτή είναι ερώτησή μου για να μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν το 7% είναι σωστό ποσοστό ή όχι. Ξεκινώ βεβαίως από την αρχή ότι τα 7% που πάνε προς το InvestEU είναι χρήμα που συνεχίζει να είναι εθνικό και τα κέρδη επιστρέφονται στα κρατη Οπότε τελικά ε, το κέρδος το, ε, αποκομί, το παίρνει το κράτος μέλος. Το InvestEU θέλουμε να είναι κάτι που θα λειτουργήσει για τους πολίτες πάνω απ' όλα εν τέλει. Ευχαριστούμε για την ΕΚΟΝ ο πρόεδρος της Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Κατάινεν που είστε εδώ. θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εξαιρετική μας συνεργασία και για αυτό το θέμα και ανυπομονώ. Εάν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα στις 25 Ιουνίου το ΕΦΣΙ γιόρτασε την, τα τρίτα του γενέθλια έχει κάτι χρονάκια πλέον. Έχει την ηλικία του αυτό το μέσο. Και θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, Αντιπρόεδρε Κατάινεν. Εάν δούμε τι χτυπήματα της μοίρα ε, είχε να αντιμετωπίσει αυτό το Εύση. και τις αποτυχίες που του ε, καταλόγησαν θα πρέπει να στραφούμε και να πούμε ότι όχι, ήταν επιτυχία, στήριξε τις επενδύσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και ήταν θετικά τα αποτελέσματά του και αυτό χάρη και στην αφοσίωση και την εντατική δουλειά του Κοινοβουλίου για να υποστηρίξει, να προωθήσει τον, ε, το έργο αυτό, το πρόγραμμα αυτό και το όλο εγχείρημα ακόμη και τι βελτιώσει του. Ευχαριστώ ιδιαίτερω του κυρίου Φερνάντε και Μπούλμαν, μάλιστα, για τη συνεισφορά του. Ωστόσο, γνωρίζουμε παρόλα αυτά ότι εάν το ΕΦΣΥ πέτυχε για να κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσει, υπολοιπόμεθα ακόμα των αποτελεσμάτων που θέλαμε να πετύχουμε, τις προσπάθειές να κινητοποιήσουμε πως, ε, αξιόλογα ποσά επιπλέον επενδύσεων για να έχουμε σταθερή ανάπτυξη και ποιότητα στα επενδυτικά έργα. Να υπάρχει δηλαδή η πραγματική, η αγνή προσθετικότητα. Ε, μας λένε οι μελέτες ότι οι επενδύσεις κάπως έχουν ε, αναθερμανθεί, αλλά βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα με τις τιμές, στις επενδύσεις των υποδομών και αλλού. Δεν έχουμε μόνο πρόβλημα με τις τιμές που δεν μπορούν να είναι στα επίπεδα της περίοδου πριν την κρίση, ούτε μόνο με την ποιότητα. Πρέπει να δούμε και τις νέες μας ανάγκες, τις νέες προκλήσεις, τις παγκοσμιοποίησεις, τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται, τις κοινωνικές συνιστώσεις. Σημαντικό και αυτό, αλλά και τα περιβαλλοντικά και τις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Υπό αυτήν την έννοια αληθεύει ότι δεν αρκεί να ε, επενούμε το ΕΦΣΙ για τις επιτυχίες του, αλλά θα πρέπει και να το ενισχύσουμε, να το προασπίσουμε, να το ε, ενδυναμώσουμε. Είναι καλή ιδέα να υπάρχει ένα νέο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εγγύηση να έχει πιο μεγάλο αντίκτυπο, να έχουμε περισσότερες δυνατότητες για επενδύσεις, περισσότερη επιλογή στους ε, εταίρους που θα συμμετάσχουν και την ανάμειξη των επενδυτικών εργαλείων. Αυτό είναι πολύ σωστό στόχος και ακριβώς ε, αυτό είναι και το ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε. Σε αυτό να προτείνουμε λύσεις. Αναγνωρίζω ότι στο κείμενο ε, βασίζεται η πρόταση στο τι έχει προηγηθεί από δουλειά ε, και στις βελτιώσεις και τις αλλαγές που μαζί ε, επιφέραμε. και πολλέ κατόπιν αιτήματο του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή μα. Υπ' αυτήν την έννοια, καλωσορίζω λοιπόν την πρόταση, αλλά θα εξετάσουμε ενδελεχώ το τι περιλαμβάνει, συζητώντα με εμπειρογνώμονε τα επόμενα βήματα τη δουλειά μα και εν γέννη ξέρω ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι. Οι στόχοι της απλούστευσης και της ευθυγράμμισης των επενδυτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα ενιαίο πλαίσιο που πράγματι θα είναι όχι απλώς ένα στοιχείο για καλύτερη διαχείριση της οικονομίας των δεξιοτήτων και την διευκόλυνση της πρόσβασης στους δικαιούχους, αλλά ταυτόχρονα η τέταρτη θηρίδα, η κοινωνική, είναι άκρο σημαντική. Μην ξεχνάμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την δυνατότητα της κοινωνικής συνοχής, τη δυνατότητα να καλύψουμε και τους ευπαθείς, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην κοινωνία. Η νέα λοιπόν αυτή, εντελώ ε, καινοτόμα και ρηξικέλευτη διάσταση θα χρησιμοποιηθεί σωστά, θα είναι αποτελεσματική αυτή η συνιστόσα θα μπορέσουμε να στρέψουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Ε, θα πρέπει να ανοίξουμε το InvestEU και σε άλλους χρηματοδοτικούς εταίρους ενδεχομένως. Πώς το βλέπετε αυτό. Θα ήθελε να μου πει ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν τι θα λέγατε σε αυτούς που ανησυχούν στο Λουξεμβούργο για τον κίνδυνο να παραγωνιστεί η ΕΤΕΠ. Η ΕΤΕΠ ε, ολοκληρώνοντας, να πω ότι μπορεί να υπάρχει μια βελτίωση ε, διαχωρίζοντα μεταξύ τη αποτυχία στην αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο εθνική αγορά ε, και την, τον κατατεμαχισμό των δύο αυτών θεμάτων. Σωστή είναι η σύνεξέταση των δύο αυτών σημείων, αλλά επειδή είπε κάποια σωστά πράγματα ο κ. Φερνάντε, να πω ότι εγώ βλέπω εδώ ένα πρόβλημα. Έχουμε μεγαλύτερη διαλεκτικότητα και ευελιξία ε, και με τα εφαρμοστικά μέτρα που δίνουμε το περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει. Όμω, αν θέλουμε περισσότερη ευελιξία, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όχι απλώς η λογοδοσία της διαφάνειας ε, θα είναι ισχυρή διάσταση, αλλά θα υπάρχει και πλήρης ε, παρακολούθηση της όλης αυτής της ε, ιστορίας από το Κοινοβούλιο και δυνατότητα να συνεισφέρει το Κοινοβούλιο. Αυτή την ευελιξία θέλουμε και αυτή την ισορροπία θέλουμε να επιδιώξουμε. Σε γενικές πάντως νομίζω ότι από εδώ μόνο στήριξη μπορείτε να έχετε για την όλη πρόταση και ακόμη και την υπόσχεση ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει πολλής χρόνος να εργαστούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος πριν το τέλος της θητείας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα είχατε την καλοσύνη τώρα να απαντήσετε στους κυρίους Φερνάντες και Γουαλτιέρη. Βεβαίως. Καταρχήν για την προσθετικότητα. Η προσθετικότητα παραμένει όπως και στο ΕΦΣΙ, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έχουμε το δημοσιονομικό κανονισμό που, που αποτρέπει την αντικατάσταση πιθανής υποστήριξης και επένδυση από άλλες πηγές της αγοράς. Αυτός είναι ο ορισμός της προσθετικότητας. Επίσης τα σχέδια, τα project θα πρέπει να τηρούν τους νέους ε, στόχους πολιτικής, να επιτυχάνουν το πολλαπλασιαστικό και μοχλευτικό αποτέλεσμα, να πολλαπλασιάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να αποτρέπουν αποτυχής αγοράς ε, και να είναι οικονομικά βιώσιμα. Η βασική διαφορά μεταξύ του InvestEU και του EFSI είναι ότι ενώ το EFSI ε, καθοδηγούνταν μόνο από τη ζήτηση, στην περίπτωση του InvestEU μας καθοδηγεί και η πολιτική, όχι μόνο η ζήτηση. Οπότε, αντί να επικεντρωνόμαστε μόνο στην ποσότητα της και την προσθετικότητα, τώρα ε, επικεντρωνόμαστε στην ποσότητα, την ποιότητα και την προσθετικότητα μας καθοδηγεί η πολιτική. Και δεν είναι ε, ίσονα σημασία αλλαγή, αλλά δεν είναι και δραστική αλλαγή. Δεν τροποποιεί ριζικά βασικά στοιχεία του ΕΦΣΥ. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς κάποιων ε, εγγυήσεων μεταξύ των παραθύρων ανάλογα με τη ζήτηση. Ε, για παράδειγμα, στο ΕΦΣΥ η ζήτηση για χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν περισσότερη από ό,τι αναμέναμε. Γι' αυτό μεταφέρθηκαν κάποιοι πόροι στο τμήμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ίδιο θα ισχύει, τέτοια δυνατότητα δηλαδή και διακριτική ευχαίρεια, θα ισχύει και με το InvestEU. Προτείναμε 15% του συνολικού πλαφών να, είναι, ε, να επιδέχεται μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τη θεματική και περιφερειακή προοπτική. Ένας από τους λόγους ε, που θελήσαμε να ανοίξουμε τον ορίζοντα πέραν του, ε, της ΕΤΕΠ, παρόλο που η ΕΤΕΠ είναι εφαρμοστικός εταίρος, γιατί έχει τη δυνατότητα ε, να δραστηριοποιείται σε όλες τις 27 ε, χώρες μέλη, γιατί 27 θα έχουν μείνει στο επόμενο πι. πι. Παρόλα αυτά, για να καλύψουμε και περιφερειακές ανάγκες, με καλύτερο τρόπο, είπαμε να ανοίξουμε τις δυνατότητες και τις εγγυήσεις και για περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την EBRD, που μερικές φορές δραστηριοποιείται περισσότερο σε κάποια κράτη-μέλη από άλλες τράπεζες. Δεν είναι ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε το μονοπόλιο της ΕΤΕΠ, που είναι και αυτός ευνόητος λόγος και εύλογος, αλλά θέλουμε να προβλέψουμε μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι να επιτρέψουμε σε αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα τις περιφερειακές ανάγκες και τους περιφερειακούς αποδέκτες από την ΕΤΕΠ να τους αφήσουμε να δραστηριοποιηθούν στη θέση της ΕΤΕΠ. Η ΕΤΕΠ ε, ε, είχε πολύ αξιόλογο έργο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και 75% ε, ε, αν μείνει τελικά, ε, είναι το ίδιο ποσό ουσιαστικά που είχε και στο ΕΦΣΥ. Εθνικά, εθνικό παράθυρο 5% είναι ήδη αρκετά υψηλό, γιατί αν δούμε ε, πόσα ταμεία συνοχής, κονδύλια συνοχής δίνουμε, σκεφτήκαμε ότι αρκούσε το 5%. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κονδύλια ειδικού σκοπού, ειδικού προορισμού για τα κράτη-μέλη που είναι πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Συνοχής για επενδυτικούς σκοπούς. Και μάλιστα συνιστώ θερμά αυτή τη ε, δυνατότητα και την αξιοποίησή της, γιατί μπορεί να έχει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τους πόρους. Τώρα, πώς συγκεκριμένα το ε, κοινωνικό παράθυρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σας έδωσα ένα παράδειγμα που προέρχεται από τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα από τις χώρες που γνωρίζω καλύτερα και που με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων έχουν ε, κάποια σχέδια κοινωνική, κοινωνικών επιπτώσεων που στόχο είναι να δώσουν θέσεις εργασίας σε 2.500 ε, μετανάστες σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις δημόσιες αρχές και με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που σας έδωσα, γιατί είναι κάτι που δεν γίνεται πολύ συχνά και είναι πραγματικά συναρπαστικό μοντέλο. Αλλά έχουμε και άλλα γνωστά παραδείγματα, όπου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΗ, έχει βοηθήσει κέντρα υγείας, επενδύσει νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Πάντως, θα πρέπει να στραφούμε ιδιαίτερος προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για τα υπόλοιπα σημεία. Η γεωγραφική ισορροπία του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΦΣΥ, ήταν ήδη αρκετά καλή. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερο δικαιούχο, δεύτερη η Εστονία, μετά η Βουλγαρία, η Πορτογαλία. Η Φιλανδία είναι η μόνη εξαίρεση. Δεν θα πρέπει ίσω να ήταν τόσο ψηλά mm. στου δικαιούχου. Μετά η Ισπανία, η Λιθουανία, Λετωνία. Οπότε το ΕΦΣΥ παρόλο που επικεντρώνεται στη ζήτηση, προσφέρει χρηματοδότηση και στις αγορές που υπέστησαν τους μεγαλύτερους περιορισμούς. Τώρα, οι λεπτομέρειες για όλα τα επενδυτικά παράθυρα θα περιληφθούν στις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις και χρειαζόμαστε κατεξοδότηση πράξη γι' αυτό και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα διαδραματίσουν το ρόλο τους αποφασίζοντας τους τομείς πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί το InvestEU. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και περάμε τώρα στους ε, σκιώδεις συγκητές. Θα ακούσουμε τους καθησυχητές των ε, ομάδων, δύο λεπτά ο καθένας και ο Αντιπρόεδρος Κατάινε θα απαντήσει αμέσως στους δύο πρώτους εισηγητές, σκιώδη εισηγητές. Πρώτη κυρία Γουαρδία Σάμπαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, μια και έχω μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή μου. Θα πάω κατευθείαν στο ψαχνό, στις ερωτήσεις. Αν και πολύ θα ήθελα να κάνω μια θετική αξιολόγηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, το InvestEU, που πολύ σωστά έχει βάλει, έχει στην στο ίδιο πλαίσιο των τριών χρηματοδοτικών μέσων και θα προσφέρει ευρωπαϊκές εγγύησεις προκειμένου να επιτύχει οικονομίες κλίμακος. Επίσης, ε, τα επενδυτικά παράθυρα είναι πολύ εύστοχη πρόταση. Πάμε σε ερωτήσεις. Το 40% για την ε, παροχή της εγγύηση. Στο πρώτο εύση είχαμε 50%, μετά μειωθήκαμε στο δεύτερο εύση το 35%, τώρα είμαστε στο 40%. Πώς καταλήξατε σε αυτό το ποσοστό, σε τι στηριχθήκατε για το 40%. Δεύτερον, περιβαλλοντική στόχη, κλιματικέ αλλαγέ. Αναφέρετε το 30% του συνολικού σχεδίου και 50% στο παράθυρο των ε, βιώσιμων υποδομών. Όταν όμως μιλούμε για βιώσιμες υποδομές, ε, πώς έχουμε 50% κλιματικές αλλαγές και το υπόλοιπο 50% σε τι θα αφιερωθεί, τι διαφορά θα υπάρχει για να διαχειριστούμε ένα ε, παράθυρο με 50% υπέρ και άλλο 50% που δεν ξέρουμε που θα δοθεί. Επίσης για την προσθετικότητα, Ρώτησε και ο κύριος Φερνάνδης και επιμένω και εγώ σε αυτό, γιατί ο ορισμός παρά είναι γενικός, πολύ πιο γενικός από ότι ε, ο ορισμός του ΕΦΣΙ για την προσθετικότητα. Και αν στο ΕΦΣΙ είχαμε σχέδια και προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν με αμφιλεγόμενη προσθετικότητα, τώρα με πιο συγκεχημένο και όριστο ορισμό, μήπως επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Επίσης, η κατανομή της εγγύησης. Ε, μας μιλήσατε για κάποια παράθυρα και κάποια καταπροσέγγιση ποσά. Σε τι στηριχτήκατε για να κάνετε την κατανομή μεταξύ τριών μεγάλων παραθύρων και ενός μικρότερου. Σε ό,τι αφορά τον κόμβο παροχή συμβουλών, το Advisory Hub, ένας από τους στόχους ε, του κέντρου αυτού είναι εντοπισμός των σχεδίων. Θα πρέπει να είναι προορατικός αυτός ο κόμβος συμβουλών. Δηλαδή, στο ΕΦΣΥ υπήρχαν κάποια προβλήματα σε αυτό το κέντρο παροχή συμβουλών. Πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε το Advisory Hub του InvestEU. Ευχαριστώ, Μέιντερ. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, τι να πρωτοπεί κανεί σε δύο λεπτά. Αυτό που με ε, εξέπληξε είναι ότι πρόκειται για κάτι καινούριο, για μια νέα πρόταση που έχει πιο πολιτικό χαρακτήρα. Για το ΕΦΣΙ 1 και 2 είχαμε κάποιο προβληματισμό. Φοβηθήκαμε ότι δεν θα είναι μεγάλη πολιτική επιρροή. Τώρα θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Αυτό όμως που δεν είναι σαφές προς το παρόν τουλάχιστον για μένα είναι ότι στο πρόγραμμα InvestEU Έχουμε ένα είδος εύση 3 συν ή είναι το εύση που κάπως αρχίζει και διαλύεται. Ποια θα είναι η νέα σχέση του InvestEU με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ερώτησή μου είναι η εξής λοιπόν. Θα θέλαμε πραγματικά αξιόλογα μέσα για να αποφύγουμε τους κινδύνους, τους χρηματοδοτικούς κινδύνους πώς ε, θα αυξήσετε τις εγγύησεις. Ε. Επίσης, ό,τι αφορά το κίνδυνο και, την, τον προορισμό των σχεδίων ή την κλίμακα των σχεδίων, έχετε περισσότερα στοιχεία. Έχουμε γιατί θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε σε πολύ ψηλέ προδιαγραφέ για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνο. Επίσης, θα έχουμε μια ένα κεντρικό διοικητικό συμβούλιο και, ένα και μια συμβουλευτική επιτροπή με έναν αρμόδιο ε, σύμβουλο επενδύσεων. Πώς θα είναι η διάρθρωση αυτών των διαφόρων δομών. Επίσης, πώς θα ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος, ο πιστοτικός κίνδυνος, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν είναι τράπεζα. Τι γίνεται με τα ιδιωτικά κεφάλαια, πώς εκτιμάτε τον αντίκτυπο των κεφαλαίων αυτών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχεδίων αν θα χρησιμοποιηθούν στο συνολικό μείγμα και ιδιωτικά κεφάλαια. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ για το 40% αυτό ε, την παροχή ήταν ε, λίγο καλύτερο το ΕΦΣΙ. Με το ΕΦΣΙ συγκεντρωνόμαστε περισσότερο σε πολιτικές όπου εκεί υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος όπως κοινωνικού τύπου επενδύσεις όπου η ε, απόσβεση δεν είναι τόσο υψηλή. Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση το καλύτερο ενδεχόμενο. Δεν θέλουμε να ενθουσιαστούμε σχετικά με το τι μπορούμε να πετύχουμε. Θέλουμε με υπεύθυνο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Αυτή είναι η όλη λογική. Ξέρετε τους αριθμούς, τα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά δεν έχω χρόνο. Ίσως αργότερα μπορώ να σας δώσω τα ακριβή στοιχεία. Προσπαθώ να καλύψω όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Γιατί 50% των υποδομών πάνε στο κλίμα. Υπάρχουν πολλές άλλες βιώσιμες επενδύσεις πέραν από εκείνες που μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακος. Κυκλικές επενδύσεις, επενδύσεις στο νερό, στην κυκλική οικονομία. Δεν μειώνουν αυτέ οι επενδύσει απαραίτητα τις εκπομπές και δεν επηρεάζει τη Συμφωνία των Παρισίων, παρόλο που είναι βιώσιμου τύπου οι επενδύσεις για βιώσιμες, βιώσιμα μέτρα. Μόνο αν υπάρχει κάτι που αντικαθιστά τους αυτοκινητόδρομους μπορεί να, υπάρχει, να θεωρηθεί σαν κάτι που περασπίζεται το, το κλίμα. Θέλουμε κάποιους ε, μελλοντοστραφεί επενδύσει, επενδύσεις, αλλά δεν μπορούν απαραίτητα αυτές να μειώνουν τις εκπομπέ. Γιατί δώσαμε 11,5 δις για βιώσιμες υποδομές, 11,5 ε, για επενδύσεις και έρευνα κοινωνικά, 4 δις. Έχουμε ιστορικά στοιχεία που κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις μας. Υπολογίσαμε πόσα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν, πώς κατανεμήθησαν και τώρα εξετάζουμε το πώς θα συναθρήσουμε τα εφιστάμενα εργαλεία. Υπάρχει κάποια προσεκτικότητα στον κοινωνικό τομέα, δεξιότητες, φερρυπίν. Αυτά που προτείναμε τα μέσα είναι σε διπλάσιο ε, όγκο. Η διαθέσιμη πόρη είναι διπλάσια από αυτούς που είχαμε μέχρι τώρα. Πολιτική επιρροή για τον κύριο Καρά. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε την πολιτική επιρροή όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων. Όχι, με τίποτα. Θέλουμε ανεξαρτησία, όπως και για το ΕΦΣΙ είχαμε αυτή την ανεξαρτησία. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατανομή των χρημάτων βασίζεται στις πολιτικές. Τα τέσσερα αυτά παράθυρα πολιτικών που σας ανέφερα. Στο ΕΦΣΙ είχαμε αναφέρει πολλούς τομείς, αλλά το ΕΦΣΙ δεν βασιζόταν τόσο στις πολιτικές αλλά σε ποσότητες, σε ποσό χρημάτων. Αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό. Συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο προηγουμένως στην επιλογή των προγραμμάτων. Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική επιρροή. Λειτουργήσε αυτό καλά και αυτή η προσέγγιση μας, μας επέτρεψε να συναθρήσουμε επενδύσεις και ο ιδιωτικό τομέας επένδυσε διότι δεν υπήρχε πολιτική παρέμβαση. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό δεν είναι ε3-0 ακριβώς, λόγω της αλλαγής προσανατολισμού. Η τεχνική υποδομή όμως ε, υποτίθεται ότι είναι ίδια. Λίγο πολύ ίδια. Η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι καλή σχέση, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι η ΕΤΕΠ δεν συμμερίζεται μαζί μας όλες τις διαστάσεις του Invest EU. δεν τους αρέσει ότι δεν υπάρχουν πλέον μονοπόλια. Το λέω αυτό, διότι ήδη θα τα ακούσατε και θα ακούσετε να αναφέρετε αυτό. Εξήγησα πριν ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι γωνιές της Ευρώπης, ακόμα και τα μικρότερα προγράμματα μπορούν να ευνοηθούν από εγγύηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα, θέλει να κάνει τα πάντα καμιά φορά κάποιες επενδυτικές ε, ε, τράπεζες τοπικές μπορεί να είναι πιο ευέλικτες και είναι καλύτερες, καλύτεροι φορείς να προωθήσουν ένα χαρτοφυλάκιο από ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση. Συζητάμε με την ΕΤΕΠ ανοιχτά τα θέματα και στο τέλος όλα θα είναι καλά για όλους. Δεν είναι τράπεζα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να είναι τράπεζα. Όλοι εκείνοι που εφαρμόζουν τα προγράμματα, Εστήθιο, EBRD, όλοι οι φορείς που εφαρμόζουν τα προγράμματα είναι αυτοί που φροντίζουν για τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς εξετάζει κατά πόσο το πρόγραμμα ταιριάζει με τις πολιτικές μας και αν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η χρηστή διαχείριση όμω και η τελική επενδυτική απόφαση εφαρμόζεται από τους διάφορους εταίρους οι συμβουλευτικές ε, υπηρεσίες και η δραστηριοποίηση. Θέλουμε οι εταίροι μας στο μέλλον να μπορούν ε, να παράσχουν ε, αυτές τις δραστηριότητες ενεργά, να δραστηριοποιούνται και ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Και τώρα, ECR, κάποιος ομιλητής από το ECR, όχι, καλώς. Άντε. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε το λόγο. Κύριε Κατάινεν, μας είπατε αρκετά από τα θετικά που είχε η αξιοποίηση του EFSI και η εμπειρία που αξιοποιείται και για το InvestEU. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αρνητικά κατά τη γνώμη σας από αυτή την εμπειρία υπήρξαν. Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα ότι χρηματοδοτήθηκαν ακριβή αυτοκινητόδρομοι στην Ολλανδία και τη Γερμανία χωρίς να υπάρχει ένας προφανής λόγος. Και προς τιμήν του και ο συνάδελφος Βανίστεν Ρόι που είναι Ολλανδός είπε «Μα δεν το φτιάξαμε το EFSI για να χρηματοδοτούμε ακριβούς δρόμους στην πλούσια Ολλανδία. Σας ε, το θέτω αυτό το ερώτημα γιατί θα πρέπει να δούμε αξιοποιώντας και τα αρνητικά από την εμπειρία πώς μπορούμε να στοχεύσουμε αποτελεσματικότερα την ενίσχυση των επενδύσεων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη αποεπένδυση, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, υψηλότερη ανεργία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο, δεν βλέπω πουθενά να αναφέρονται κοινωνικοί δείκτες στα κριτήρια με τα οποία θα λαμβάνονται τελικά οι αποφάσεις για το πού θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις, όπως μακροχρόνια ανεργία, νεανική ανεργία, ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σας απασχολεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να βάλετε και κοινωνικά κριτήρια. Και μια δεύτερη ερώτηση υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κατηγορούνται, ελέγχονται και ορισμένες έχουν καταδικαστεί κιόλας, έχουν υποστεί κυρώσεις για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Σκοπεύεται εταιρείε που βαρύνονται με τέτοιες παρανομίες να τις αποκλείεται από τη συμμετοχή σε τέτοιες επενδύσεις. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν για την παρουσίαση. Πρέπει να πω ότι στο παρελθόν είχαμε επικρίνει δρυμιαίο στο. ε, ΕΦΣΥ επειδή θα μπορούσε υποτίθεται να αναθερμάνει μόνο τη ζήτηση αυτό σε κάποιες συγκεκριμένε χώρες. Παρόλα αυτά, με την δεσμευτική προσθετικότητα που ήταν απαραίτητη, περάσαμε γρήγορα από το FC1 που δεν προέβλεπε αρκετή προσθετικότητα στο 2 που ήταν αυστηρότερο αυστηρότερο. Οπότε υπήρχε και κοινωνική διάσταση και άλλες προεκτάσεις που μας απασχολούσαν. Πάντως, αυτά τα 650 υποθετικά δις θα έχουν έναν αντίκτυπο αρκετά μακροπρόθεσμο, διότι με την ε, διέρεση στα 7 χρόνια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και τα 27 κράτη-μέλη, τελικά δεν είναι και τεράστιο το ποσό αν το διαιρέσει κανείς. Πάντως, εκτιμώ την πρόταση που έχετε κάνει να προβλεφθεί στην εγγύηση του Invest EU να πάει εκεί ένα μέρος των διευθυντικών κονδυλίων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και μετά τα κονδύλια αυτά, αφού συγκεντρωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ανακατευθυνθούν προς το κάτω μέλος. Ε, αυτό βέβαια πρέπει να δούμε ε, και να, αν μπορεί να διευκρινιστεί περαιτέρω για να ξέρουμε τι δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες. Διότι υπάρχει, υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ευχαρίστως. Ευχαριστούμε και τώρα στη δικασία Catch ο κύριος Σαρβάμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, με συγχωρείτε, πρώτα πρέπει να έχουμε τις απαντήσεις γιατί ήταν δύο οι ερωτήσεις. Δύο οι ερωτώντες. Πρώτα η απαντήση του κ. είναι μετά το Κατστιαί. Ευχαριστώ πολύ. Για τους ακριβούς αυτοκινητοδρόμους. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο ακριβή, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει αρκετά αυστηρούς κανόνες για την χρησιμοποίηση του ΕΦΣΙ 2,0 για αυτοκινητοδρόμους. Δεν βλέπαμε να έχει νόημα. Υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις. για κάποιες χώρες συνοχής ή τη διασύνδεση κάποιων χωρών συνοχής με κάποιες άλλες. Η πρότασή μας δεν πέρασε όσο είχε λόγω του και κάποιων άλλων αποφάσεων των συνομοθετών. Αλλά το ΕΦΣΙ δεν χρηματοδοτεί, ε, ούτε πρημοδοτεί τέτοια ακριβά έργα όπως το αυτοκινητόδρομοι. Ενδεχόμενες αρνητικές πτυχές και συνέπειες του Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας ε, σοβαρός κίνδυνος που έχει προκύψει από τις ε, εκτιμήσεις μας και τις αναλύσεις μας κίνδυνος ε, σε σχέση με την προσθετικότητα. Δηλαδή, ε, ο κίνδυνος των, ιδιωτικών, των ιδιωτών επενδυτών να ε, βγει εκτός του παιχνιδιού. Ουσιαστικά δηλαδή να την πληρώσουν οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν χρειάζεται να την πληρώνουν, μάλλον ε, το αντίθετο. Οι ιδιωτικοί επενδυτέ, οι ιδιώτε επενδυτέ να μην πάρουν αρκετά μέρο. Δεν χρειάζεται τα λεφτά, τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται αντί για τον ιδιωτικό τομέα. Οι εταιρείε τώρα που είχαν προβλήματα με την δικαιοσύνη, όντως είχαν μπει σε μαύρη λίστα. Είναι σωστό αυτό που είπατε λοιπόν. και το τμήμα της χρηματοδότησης από κάτι μέλη προς το Invest EU. Είναι καινοτομία αυτό, είναι μια, ε, ένας νεοτερισμός. Τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν το επιπλέον 5% των ε, διευθυντικών ταμείων να τα πάνε σε κάποια από, σε κάποια τις που έχουμε προβλέψει. Ε, ας πούμε τις δεξιότητες και κάποιες κοινωνικές διαστάσεις, τις κοινωνικές επενδύσεις. μπορούν να πάρουν τη συνολική μόχλευση του InvestEU μετά για να τη χρησιμοποιήσουν στη χώρα τους για αυτό το σκοπό. Εάν τελικώς δεν χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα που διατέθηκαν, θα επιστραφούν στο κάτω μέλος. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα εδώ. Η μόχλευση είναι πολύ μεγαλύτερη στο σύνολο παρά για το καθένα από τα κράτη-μέλη μόνο του. Και μπορεί όντω να λειτουργήσει ω καταλήτη για τι ιδιωτικέ επενδύσει. Ελπίζουμε ότι οι συνομοθέτε, ο θα το, οι συνομοθέτε μάλλον θα το δεχτούν αυτό. Και ότι το μήνυμα θα περάσει. Διότι σε ορισμένα κάτι μέλη μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Για τον κοινωνικό αντίκτυπο αναφέρεται ξεκάθαρα στην ε, θηρίδα, στο παράθυρο των ε, κοινωνικών ε, υποδομών. Είναι κάτι που λέγεται ξεκάθαρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Σαββάρμα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο Κατάιναν, γιατί πραγματικά προσπαθεί εργοδός να ενισχύσει κάτι που έχουμε ήδη, γιατί υπήρξαν πολλές αμφιβολίες και επικρίσεις για το ΕΦΣΥ και είχα το προνόμιο να συμβάλλω στο ΕΦΣΥ δεύτερης γενιάς στον τριμερή διάλογο και ε, έριξα μια πιο διεξοδική ματιά σε αυτό και είναι καλή αυτή η προσπάθεια να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό έχω και κάποια σχόλια για να συμβάλλω και εγώ στην περαιτέρω βελτίωση. Καταρχήν, οι ανησυχίε από την προοπτική του ορίζοντα, του προγράμματο ορίζοντας, ε, ότι δηλαδή θα ε, χαθούν κονδύλια από τον ορίζοντα, ιδιαίτερα για τη βασική έρευνα πώς θα διασκεδάσετε αυτές τις ανησυχίες. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Κάρας, όντως ε, το InvestEU ναι μεν θα κατευθύνεται περισσότερο από την πολιτική, αλλά θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της οικονομικής βιωσιμότητας των σχεδίων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φερνάντες, Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Εγώ πιστεύω ότι και το πρώτο και το δεύτερο εύση ξεκίνησαν για να ε, γεφυρώσουν το επενδυτικό κενό που προκάλεσε η κρίση στην Ευρωζώνη. Πολύ ε, σκεφτήκαμε ότι χρειαζόμαστε ένα αντικυκλικό μηχανισμό που με κάποια κρατική δημόσια βοήθεια θα αναζωογονούσε την εθνική ζήτηση εν μέσω της κρίσης. Το θέμα είναι ότι Μερικές φορές φαίνεται ότι οι μηχανισμοί ε, αυτοδικαιολογούνται. Υπάρχει κάποιο αντικυκλικό στοιχείο στη δική σας τελευταία πρόταση. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι υπάρχει άλλος ε, κανονισμός για τον αντικυκλικό μηχανισμό της Ευρωζώνης και ισχύει αυτό. Αλλά αν όμως χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές συνοχής, να βελτιώσουμε τις μεταφορές, τις υποδομές μας, δεν θα ήταν καλύτερο να συμβάλλουμε με περισσότερα κονδύλια στον κοινοτικό προπολογισμό, στον ενωσιακό προπολογισμό ή στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί αν θέλουμε έναν αντικυκλικό μηχανισμό, δεν ξέρω σε τι βαθμό μέχρι ότου έχουμε στο μέλλον αυτόν τον κανονισμό, γιατί τώρα ξεκινάνε οι επενδύσει, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να χάσουμε την ικανότητα που μα έχει δώσει αυτό ο μηχανισμό να δούμε ποιο είναι ο βαθμός μόχλευση ετησίω των προγραμμάτων για να δούμε ποιο είναι το επενδυτικό κενό. Δεν θα πρέπει, πιστεύω, να χάσουμε και αυτή την ε, πτυχή. Ευχαριστώ. Κύριος Βανίλ Ρόι. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις. Εγώ είμαι μέλος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και εκεί θα συντάξουμε γνωμοδότηση για το πρόγραμμα και μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα συμφωνήσουμε για το πακέτο Omnibus και στο πακέτο αυτό εξετάσαμε μέσα σαν το ΕΦΣΙ και το πρόγραμμα InvestEU και είπαμε ότι ε, τα χρήματα που βρίσκονται στα εθνικά, ε, στα εθνικά προγράμματα δεν θα πρέπει να πάνε σε να γυρίσουν στην Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν ε, σε προγράμματα όπως το EU Invest ή το EFSI. Γιατί είπατε ότι τα χρήματα θα πάνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστρέψουν στα κράτη-μέλη. Ερωτώ λοιπόν. Αν, είμαστε, αν συνεργαζόμαστε κατευθείαν με τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες, στην Ολλανδία έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί χρειάζεται να φέρουμε πρώτα τα κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν να μην χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς μέσω των περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. Γιατί να βγάλουμε τα χρήματα αυτά από τους εθνικούς φακέλους. Συμφωνώ με το 5% αλλά είναι πιο τεχνική η ερώτησή μου. Γιατί την επόμενη πέμπτη θα αποφασίσουμε αν είναι ε, απαραίτητο στο γενικό κανονισμό. Ο Αντιπρόεδρος Κατάιναν. Ευχαριστώ για το θέμα του προγράμματος Ορίζοντας. Ευχαριστούμε κύριε Σαβερμά που το αναφέρατε, γιατί άκουσα και εγώ κάποιες αφιβολίες ή κάποιες ανησυχίες ότι πάλι η Επιτροπή ε, κλέβει από το Ορίζοντας. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν βάζουμε χέρι στο πρόγραμμα Ορίζοντας. Όταν μιλούμε για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, είναι ότι χρησιμοποίησαμε χρηματοδοτικά μέσα του και συνδυάσαμε χρηματοδοτικά μέσα του ορίζοντας 2000 που πηγαίνουν μέσα στο InvestEU και έχουν ε, αφιερωθεί για ε, ειδικό προορισμό, την έρευνα και την καινοτομία. Και με την κοινή συγκέντρωση, το pooling, θα αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στην έρευνα και την ε, καινοτομία. Και τα κονδύλια αυτά ούτε στον ορίζοντα 2000 πήγαιναν στη βασική έρευνα. Γιατί δεν, μπορού, δεν μπορεί κανείς να πάρει δάνειο για να πληρώσει μισθούς. Για το μετοχικό κεφάλαιο της Ινοφίν και η Ινοφίν χρησιμοποίησε άλλα σχέδια έρευνας και καινοτομίας. Η ιδέα θα παραμείνει ως έχει σε μεγάλο βαθμό, αλλά ο όγκος συνολικός θα αλλάξει γιατί με μεγαλύτερη κλίμακα θα χρηματοδοτήσουμε περισσότερα καινοτόμα και ερευνητικά σχέδια. Αλλά και το παράθυρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τα καινοτόμα σχέδια και προγράμματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και πάλι δεν θα έχουμε ε, πολιτική παρέμβαση στην επιλογή των προγραμμάτων. Δεν θα υπάρχει πολιτική επιρροή, γιατί αυτή η αρχή της ανεξαρτησίας λειτουργεί καλά γιατί προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ιδιωτικά κεφάλαια και να τα συνδυάσουμε με το ΕΦΣΥ. Δεν θέλουμε επουδενή να καταστρέψουμε ένα σύστημα και ένα μηχανισμό που λειτουργεί καλά στο ΕΦΣΥ. Τώρα για τον αντικυκλικό χαρακτήρα του EFSI, του και το αν θα πρέπει να μεταφερθούν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κονδύλια. Και ναι και όχι. Όχι με την έννοια ότι αν θέλαμε να κάνουμε κάτι αντικυκλικό, θα έπρεπε να μειώσουμε τις επενδύσεις. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν ανάγκες πολιτικής, για παράδειγμα η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, ή υπάρχει ανάγκη σε επενδύσεων σε κοινωνικές υποδομές, σε δεξιότητες, σε καινοτομία και έρευνα, Γι' αυτό και το InvestEU δεν είναι μόνο αντικυκλικό, αλλά είναι και ε, πυροδοτή πολιτική ουσιαστικά. Επίσης, η προσθετικότητα εξακολουθεί να έχει τη σημασία της. Δεν θέλουμε να εκτοπίσουμε τα ιδιωτικά κονδύλια, τις ιδιωτικές επενδύσεις. και έτσι προστιθέμεθα σε αυτά που κάνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είπατε γιατί να μην αυξήσουμε το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕΠ για να ενισχύσει περισσότερες δράσεις ή να αυξήσουμε τον ενωσιακό προϋπολογισμό ή να έχουμε έτσι περισσότερους πόρους στο Ταμείο Συνοχής. Η διαφορά μεταξύ InvestEU και των άλλων δύο προτάσεων είναι ότι τα κονδύλια της συνοχής είναι επιδοτήσεις ένα εκατομμύριο επιδοτήσει στην συνοχή δεν έχουν καμία μόχλευση. Ένα εκατομμύριο παραμένει ένα εκατομμύριο. Αν όμω χρησιμοποιήσουμε ένα εκατομμύριο ω κεφάλαιο ή εγγύηση, τότε έχει μεγαλύτερη μόχλευση. Χρειαζόμαστε λοιπόν και επιδο... επιδοτήσει από τη μια πλευρά και χρηματοδοτικά μέσα από την άλλη. Για να προσελκύσουμε και ιδιωτικά και δημόσια κονδύλια. Οι επιδοτήσει δεν αρκούν για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕΠ, αυτό θα το αποφασίσουν τα μέλη της ΕΤΕΠ, θέλουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και πάλι εδώ ε, το InvestEU έχει προστιθέμενη αξία, γιατί αφήνει, ε, ανοίγει τις εγγύησεις και σε άλλους εταίρους, όχι μόνο στην ΕΤΕΠ. Μερικές φορές και περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες είναι πιο ευέλικτες για να κάνουν τη δουλειά που δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει η ΕΤΕΠ. Εξού και η προστιθέμενη αξία του InvestEU στο άνοιγμα των εταίρων και προς περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Επίσης, το Εθνικό Κονδύλιο είναι ε, προαιρετικό. Φυσικά οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν όσο και όπως μπορούν. Αλλά αυτό είναι σε θελοντική βάση, προαιρετικό. Σε πολλέ περιπτώσει, το τριπλό α τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ θετικό και προσελκύει κεφάλαια. Είναι πολύ σημαντικός παράγον αυτή η θετική αξιολόγηση του τριπλό α τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θέλουμε να θεωρούμε τα κράτη-μέλη να δουν τι ευκαιρίε δίνουν τα χρηματοδοτικά μέσα και πέραν της ε, χρηματοδότηση της συνοχή που εδράζεται μόνο σε επιδοτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ήταν χρησιμότατη και πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που έλαβε χώρα. Έχουν περισσότερα στοιχεία για την έναρξη του νομοθετικού μας έργου το οποίο νομοθετικό έργο θα προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν και όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και για την ποιότητα της ε, προτάσεως αυτής. Προσβλέπουμε σε καρποφόρα συνεργασία στο θέμα αυτό. Ζων, θες να πεις κάτι, να προσθέσεις. Σας ευχηθώ καλό βράδυ και να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι ένας νέος μοχλός ανάπτυξης αυτό το μέσο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.